Σας καλωσορίζω. Πρόκειται για την τελευταία συναντρία της Επιτροπής μας για φέτος. Μετά θα συνεχίσουμε βέβαια, αλλά και φέτος είναι τελευταία. Προσωρινή ημερήσια διάταξη έχετε λάβει, υπάρχουν αντιρρήσεις. Όχι, εγκρίνεται επομένω. Πρακτικά 13 Οκτωβρίου, 3 4 Νοεμβρίου υπάρχουν ε, προβλήματα εδώ, οι δάλος εγκρίνονται. Και θα ήθελα να επισημάνω ότι αύριο στις 12, μια και είναι η τελευταία συνεδρίαση της ε, χρονιάς, θα κάνουμε μια μικρή γιορτή και τα Χριστούγεννα. Ένα ποτό. Και σας προσκαλούμε όλους. Σημείο 4 στην ημερήσια διάταξη. Παρουσίαση της Επιτροπής για το ε, νέα έκδοση του προγράμματος εργασίας και του πακέτου εργασίας για το μέσο συνδέοντας στην Ευρώπη 2014. Ο κύριος Ονίλη είναι εδώ εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει 15 λεπτά στη θέση του για να μας παρουσιάσει το πρόγραμμα και να ακολουθήσει η συζήτηση. Κύριε Ονίλη, έχετε το λόγο παρακαλώ.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 legal base was adopted by you, we had to conduct an ex ante study. This ex ante study has been uh, και έπρεπε να κάνουμε μελέτη εκ των προτέρων και άρα ήταν σοφό να ξεκινήσουμε με ένα εργαλείο το οποίο να είναι εργαλείο ε, ε, δανείου χρέους, debt instrument και όχι εργαλείο ίδιων κεφαλαίων, equity. Και έχουμε τέτοιες δυνατότητες ε, περαιτέρω ε, πίστοσης ε, σε αυτούς που θα αναλάβουν όλα αυτά τα project. Τα ποσά λοιπόν είναι τα εξής. Έχουμε 127 εκατομμύρια ευρώ από αυτά ο κλάδος των μεταφορών θα πάρει τη μερίδα του λέοντος 70 εκατομμύρια, 60,5 εκατομμύρια ευρώ για τηλεπικοινωνίες και σχεδόν 41 εκατομμύρια για την ενέργεια. Αυτά τα εργαλεία θα τα διαχειριστεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα γίνει ε, συμβατική ρύθμιση έτσι ώστε να εφαρμόσει αυτούς τους μηχανισμούς, αυτά τα εργαλεία. Σκοπός είναι να προωθήσουμε δύο κατηγορίες ε, project, πρωτοβουλίες με ομόλογα έργου, τις οποίες ίσως γνωρίζετε αρκετά καλά, project bond, αλλά και άλλες ε, δυνατότητες πίστοσης και εγγυήσεων. Αυτό θα γίνει κατόπιν συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και θα έχουμε τη δυνατότητα και του χρόνου να συναντηθούμε με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για να σας παρουσιάσουμε τα είδη των έργων που δρομολογούνται και που μπορούν να είναι επιλέξιμα. Οι δυνατότητες λοιπόν που είναι διαθέσιμες από την αρχή της επόμενης χρονιάς θα είναι και το εργαλείο άμας για να προωθήσουμε νέα έργα μέσω πίστοση και εγγύησεων. Οι προτεραιότητες είναι ίδιες, δεν έχει αλλάξει κάτι. Οι προτεραιότητες είναι αυτές που έχετε εσείς απαριθμίσει. Έργα που εξυπηρετούν τους διάφορους διαδρόμους, corridor και σε διάφορους τομείς. Ε, ε, Υδάτινοι δρόμοι εσωτερική, λιμένες μεταξύ άλλων. Με αυτό το μηχανισμό δανεισμού πίστοσης ε, εξετάζουμε το ενδεχόμενο να έχουμε συγκεκριμένα έργα για συγκεκριμένους θεματικούς άξονες και ελπίζουμε στα, μέσα της ε, επόμενης χρονιάς να είμαστε σε θέση να περιγράψουμε πολύ συγκεκριμένα εργαλεία για το ERTMS και για την περαιτέρω ενθάρρυνση του ΣΕΣΑΡ που είναι για ε, την αεροπορία για την χρηματοδότηση επίσης καθαρών δημόσιων μεταφορών έτσι ώστε οι μεγάλοι δήμοι να μπορούν να αξιοποιήσουν αυτές τις δυνατότητες ε, χρηματοδότησης για να επενδύσουν σε νέες δημόσιες μεταφορές πολύ πιο καθαρές. Και ελπίζουμε να έχουμε ε, νέο ταμείο μεταφορών για να εξυγχρονίσουμε τις ε, υδάτινες ε, οδούς μεταφορών στο εσωτερικό. με καθαρότερους κινητήρες και καλύτερα συστήματα πληροφόρησης. Δεν υπάρχει άμεση σχέση με την πρωτοβουλία, ε, την χρηματοδοτική που σας παρουσίασε ο πρόεδρος κ. Γιούνκερ την περασμένη εβδομάδα. Είναι τελείως διαφορετικά τα μεγέθη αλλά είναι και τελείως διαφορετική η ουσία αυτών των ε, μέσων. Θα είμαι εξαιρετικό, εξαιρετικά σύντομος, γιατί νομίζω ότι η Επίτροπος Bulk, ε, Βιολέτα, θα έρθει αύριο και θα σας παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιηθεί καλύτερα αυτό το οικονομικό μέσο. Θέλω όμως να πω ότι Αυτά που συζητούμε εδώ θα είναι διαθέσιμα από την αρχή της επόμενης χρονιάς. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε μέχρι τα μέσα αυτής της χρονιάς. Και θα χρησιμοποιηθούν για συγκεκριμένα έργα, π.χ. εξυγχρονισμός και επέκταση του λιμένα του Καλέ ή κατασκευαστικές εργασίες στο έργο του Άμστερνταμ ε, για την ε, ε, καταπολέμηση της ροής των υδάτων και, την, και τα φράγματα εκεί που είναι απαραίτητα, μεταξύ άλλων. Βλέπετε ότι Έχουμε πάρει την απόφαση να ε, έχουμε μικρότερα μέσα, τα οποία όμως να αλληλοσυμπληρώνονται. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Για να δούμε τους συντονιστές πρώτα, αν έχουν κάτι να πούν. Κύριος Φαντεν Κάμπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Ήταν σαφής. Και αυτό που δεν έχω καταλάβει είναι για ποια χρονιά προβλέπεται η δαπάνη των κονδυλίων. Από αυτά που άκουσα εγώ τώρα βγάζω συμπέρασμα ότι είναι για το 2015. Το μέσον συνδέοντας την Ευρώπη είναι νέο, αλλά βλέπω ότι τα ποσά γράφονται ήδη για το 2014. Ποιος είναι ο σχετισμός εδώ. Πρέπει να περιμένουμε μέχρι να έρθει η κυρία Βουλσάβρου να μας μιλήσει. Με το σχέδιο του κυρίου Γιούνκερ. Ξέρουμε όμως ότι ο κύριος Γιούνκερ έχει αφαιρέσει ποσά από το Connecting Europe. Επομένως, τι θα βγει τελικά. Τα 17 από εκατομμύρια είναι μεγάλο ποσό. Ο πρόεδρος, ευχαριστώ. Ισμαήλ Ερτού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον κύριο Νιντή για την ε, παρουσίαση. Έχω δύο ερωτήσεις, το προσπαθώ να τις συνοψίσω σε μία. Αν κατάλαβα καλά, λόγω των δυσχεριών που παρουσίασε η αγορά, θα το πούμε, ε, αναζητήθηκαν ε, διαφορετικά μέσα, εναλλακτικέ. Με αυτό το μέσο αφενός με δανεισμού και αφετέρου των ιδίων κεφαλαίων, το equity. Ε, συγκεκριμένα όμως τι θέλετε να πείτε. Αυτό το μέσο ιδίων κεφαλαίων θα τεθεί σε εφαρμογή σε μια δεύτερη φάση. και άρα θα ε, τύχει διαχειρίσω σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Συγκεκριμένα αυτό πώς προβλέπετε να γίνει, γιατί όταν είχα εγώ την ε, ε, έκθεση ως εισηγητής για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, βρισκόμουν πάντα αντιμέτωπος με μια ερώτηση. Τι, μου, τι σημαίνει για μένα αυτή η νομοθεσία, εμένα τον επενδυτή, τον επίδοξο επενδυτή. Τι θα πρέπει να απαντήσουμε λοιπόν εδώ έρχεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και αναλαμβάνει μέσω εγγυήσεων επαραδείγματι εμπράγματων ενδεχομένως την ε, απρόσκοπτη λειτουργία του προγράμματος ώστε να μπορούν να μπουν μέσα οι επενδυτές. Εάν η απάντηση είναι καταφατική μου αρκεί ένα ναι. Εάν όχι χρειάζεται πες εξηγήσει. Γιατί εδώ όταν μιλούμε για η ίδια κεφάλαια χρειάζεται να υπάρχουν τα κεφάλαια αυτά. Χρειάζεται να έχουμε στη θέση μας το χρήμα αυτό και να ξέρουμε και πώς θα το διαθέσουμε. Αν λοιπόν εδώ πέρα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων διαθέτει μόνο ε, τις εγγύησει, τότε μου αρκεί μόνο ένα ναι. ή Ιδάλλως χρειάζομαι πιο πολλές εξηγήσεις. Ευχαριστώ κύριος zullen zeker met eh, de commissaris morgen nog eens even precies inzoomen op de financiële consequenties. Eh, dat doen we morgen. Σας ευχαριστώ. Σίγουρα θα συζητήσουμε αύριο το πρωί τις οικονομικές συνέπειες, αλλά εγώ θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία σήμερα. Ο κύριος Νίντι μίλησε για την ε, νέα αποβάθρα στο Άμστερνταμ. Και θα ήθελα να καλέσω όλους σε Μία από τις αίθουσες στις 6.30 θα γίνει παρουσίαση για τη συγκεκριμένη ε, αποβάθρα και θα σας δω απόψε στην ε, συνάντησή μας. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ήταν προγραμματισμένο αυτό, αλλά καλές είναι οι εκπλήξεις. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρον. Και καταρχάς ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Όντως, πάντα με χαρά βλέπουμε να υπάρχουν διαθέσιμα στον τομέα των μεταφορών τουλάχιστον χρήματα, αλλά τα ερωτήματα αναπόφευκτα δεν τυπώνονται. Πόθεν θα έρθουν τα χρήματα αυτά και πώς θα συνδεθούν μέσα στο Connecting Europe. Γιατί ξέρουμε τα λεφτά μόνο μια φορά που θα τα δώσουμε. Ξέρουμε τι έχει προκύψει με τον προϋπολογισμό. όπως συμφωνήθηκε το, στο τέλος του προηγούμενου έτους η ιστορία με το Connecting Europe. Ε, να πολλαπλασιάσουμε το χρήμα δεν γίνεται, ιδάλλως θα το είχαμε κάνει όλοι και τώρα πρέπει, τουλάχιστον αυτό ζητούν και τα κράτη-μέλη, εάν θέλει κανείς να χρηματοδοτήσει μετά το 2015 ένα έργο, να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που υπάρχουν, σαν αναφερθήκατε σε έργα όπως ο Λιμένας του Καλέ ή του Αμστερντάμ, που προχωρούν με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν λοιπόν και άλλα κράτη-μέλη που έχουν διατυπώσει σχετικό αίτημα και αν κάποιοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να βιαστούν γιατί τα χρήματα τελειώνουν. Ναι. Δεύτερη ερώτηση. Ένα πρόσθετο πακέτο το οποίο ενδεχομένω να προκύψει θα πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες του συνδέοντας την Ευρώπη ε, θα υπάρχουν επιλογές για τη χρηματοδότηση οδικών δικτύων ε, ενδεχομένως ή πάντα μένουμε στον περιορισμό των θαλασσίων και των σιδηροδρομικών μεταφορών. Ε, γιατί δεν είναι σαφές για μένα. Ευχαριστώ κυρία Κίλεν. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι σαφές ότι οι στόχοι είναι εξαιρετικά φιλόδοξοι. Όλοι μας θέλουμε να τους επιτύχουμε. Όμως σε μένα με ανησυχεί η κατάσταση, διότι για κάθε πρόγραμμα έχουμε ε, και ένα μεγάλο κομμάτι εθνικής χρηματοδότησης. Εδώ λοιπόν δεν μιλάμε μόνο για ε, ευρωπαϊκά κονδύλια αλλά και για εθνικά κονδύλια. Δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα. Θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες αξιολογήσεις ε, όσον αφορά την εθνική συμμετοχή κάθε φορά. Πώς έχει υπολογιστεί ή μήπως περιμένουμε τον Άγιο Βασίλη να έρθει και να μας τα χαρίσει. Ε, ναι, αλλά πρώτα έρχεται ο Σαν Νικολά, ξέρετε, 6 Δεκεμβρίου και μετά ο Άγιος Βασίλης. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Η κυρία Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση αυτή. Εγώ έχω πολλές ερωτήσεις. Καταρχήν αυτά τα μέγα έργα, είτε είναι η Λιόν είτε είναι το Μπρένερο, Θέλω να ξέρω το εξή σε ποιο βαθμό θα λάβουν κονδύλια ευρωπαϊκά, ποιο είναι το ακριβές ποσοστό. Πρέπει να μας δώσετε στοιχεία. Εδώ λέτε ότι πρόκειται για μια αξιολόγηση για ένα προσχέδιο χρηματοδότησης, άρα λοιπόν το πραγματικό πρόγραμμα εργασίας θα έρθει προσεχώς. Ερώτηση. Υπάρχει λοιπόν προσέγγιση για το πώς θα συμπεριληφθεί η πρωτοβουλία των τριών δις του κυρίου Γιούγκερ μέσα σε αυτές τις ε, δημοσιονομικές, ε, δημοσιονομικό πραγματισμό. Δεύτερον, πώς το θέμα του ελλείμματος αντιστοιχεί με τους στόχους ε, της, της Κομισιόν για να μπορέσουν τα κατημέλη να μειώσουν το χρέος τους. Και μια τρίτη ερώτηση έτσι μόνο και μόνο για τη χαρά να θέσει αυτή την ερώτηση είναι θέλω να ξέρω γιατί η Κομισιόν ελπίζει πως οι ιδιωτικέ επενδύσεις, ενώ για την ώρα δεν έχουμε πραγματικά στοιχεία που να δείχνουν ε, κάποια επιτυχία, γιατί η Κομισιόν ελπίζει πως αυτές οι ιδιωτικές επενδύσεις μπορεί να ενδιαφέρουν για μακροχρόνιες δεσμεύσεις και δανεισμό στις υποδομές των μεταφορών. Μπορώ να έχω απαντήσεις από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Τζιλ Σάιμον. Σαϊμούρ. Σαϊμούρ. Nicht da? Dann kommt Monsieur Riquet. Merci, Monsieur le Président. Ο κύριος Ρικέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλά τα ερωτήματα που θα ήθελα να θέσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα μπορέσω να τα θέσω όλα και γι' αυτό θα περιοριστώ σε πολύ λίγα. Για παράδειγμα, για ε, τα χρηματοδοτικά μέσα. Δεν θα μιλήσω για τα, την επιλογή των έργων, αλλά για το θέμα του, του πώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός. Πρώτον, λοιπόν, τα έργα στα οποία αναφερθήκατε είναι αυτά για τα οποία έχει υποβληθεί πρόταση στην ε, πρόσκληση υποβολής προτάσεων έργων του Φεβρουαρίου του 2015, 14, με συγχωρείτε, είναι μέσα σε αυτά ή είναι άλλα. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Δεύτερο, σε σχέση με τα ομόλογα έργου και τις προθεσμίες, με τη μελέτη εκ των προτέρων και τη μελέτη εκ των, προ... υστέρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τι θα συμβεί ε, σε αυτό το χρονικό διάστημα που θα έχει ολοκληρωθεί η, κατανομή των κονδυλίων μέχρι ότου να ολοκληρωθεί και η μελέτη. Τρίτο ερώτημα, το εξής. Με δεδομένη τη θέση του Συμβουλίου για αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα, εξαιρετικά επιφυλακτική. Ανέκαθεν η θέση του Συμβουλίου, το οποίο ανέκαθεν προσπαθούσε να περιορίσει την αξιοποίηση αυτών των νέων ε, χρηματοδοτικών μέσων και των ε, καταληκτικών, αν θέλετε, ποσοστών. Μπορεί να τροποποιηθεί αυτή η πρότασή σας με αυτό το δεδομένο. Γιατί με εξέπληξε το γεγονός ότι το πρόγραμμα Juncker βασίζεται στο ότι τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία θα λειτουργήσουν ως μοχλός πίεσης, ενώ το Συμβούλιο ήταν ε, πολύ εναντίον αυτών των δυνατοτήτων. Ε, προσιλητίστηκε το Συμβούλιο ξαφνικά ε, και τα επιθυμεί πλέον. Και τέταρτη και τελευταία ερώτηση εξή. Δεδομένου του γεγονότος ότι βάσει του σχεδίου Juncker προβλέπεται να έχουμε 3,2 δις στο μηχανισμό συνδέοντας την Ευρώπη, θα αναθεωρηθεί η νομική βάση. Αυτό το θεωρώ απαραίτητο. Υπό ποια έννοια και μέχρι πότε και με βάση ποιου χρονοδιαγράμματος. Και, συν της άλλης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει ε, αν αυτά τα 3,2 δις θα παρθούν από το φάκελο των 33 δις ή από το φάκελο για την ανταγωνιστικότητα ή από πού θα ε, έρθουν αυτά τα 3,2 ε, δις αναλόγως με, την, με τον τομέα που μας απασχολεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Γιάννη Συνέλης είναι τελευταίος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω κάποια σκέψη εδώ. Πριν από μερικές εβδομάδες λάβαμε μια έκθεση ανέθεσε το Κοινοβούλιο μια μελέτη ε, που αφορούσε τους μεγάλους διαδρόμους. Με την έκθεση λοιπόν αυτήν, στην οποία συνεργάστηκε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διατυπώθηκαν καλές συστάσεις από ό,τι υπόθηκε, εκ των οποίων η μία έλεγε ότι θα πρέπει να μεριμνήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμη περισσότερο να προκαταβάλει, ε, front loading δηλαδή, ε, τις, ε, διορθώσεις σε σχέση με τους διαδρόμους. Αυτό μπαίνει τώρα μέσα στο πρόγραμμα εργασίας. Ευχαριστώ, Φαντανκάμπ. Ναι, Πρόεδρε, ε, ζητώ συγγνώμη γιατί ξέχασα τελείως μια σημαντική, πολύ σημαντική ερώτηση. Έγινε λόγος για το EMTS και την ε, ανακαίνιση στο χώρο των σιδηροδρομικών μεταφορών. Αυτό ισχύει όμως και για τις εσωτερικές φλωτές συγκοινωνίας, γιατί έχουμε εκεί πολλά σκάφη τα οποία θα μπορούσαν ε, να ανακαινιστούν, να αναδιαμορφωθούν και αυτό θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορεί να υπαχθεί στο σύστημα του συνδέοντα στην Ευρώπη. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Θέλω και εγώ να κάνω μια ερώτηση. Αν υπάρχει τρόπος ε, κάπου μέσα από το Connecting Europe να ε, χρηματοδοτηθούν έργα που χρειάζονται ε, ανακαίνιση, διόρθωση και που δεν έχουν καθόλου αξιοποιηθεί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επίσης για τη χρηματοδότηση που έγινε λόγος, γιατί έμαθα ότι για τους κύριους διαδρόμους της Ευρώπης και ο κυριότερος είναι Ρότερνταμ-Γενέβη γίνεται στην Ιταλία ακόμη η ανέγερση, η εγκατάσταση μάλλον των στοδρομικών γραμμών. Οι Ελβετοί μου λένε «Α, εμείς ε, φτιάχνουμε το δικό μας κομμάτι, αλλά με δική μας χρηματοδότηση». Οι Ιταλοί όπου να είναι ξεκινάνε. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, σε καμιά 33 χρόνια θα έχουμε κανένα 15% του έργου έτοιμο. Ε, εσείς σε αυτό τι έχετε να πείτε, σας αρκεί να λέτε ότι προχωράει ο καθένας από την πλευρά του αργά-αργά, γιατί η Ιταλία δεν έχουν κάνει, οι δεν έχουν κάνει τίποτα και ούτε και οι Γερμανοί πρέπει να πω. Ή αλλιώς θα πείτε, μια και η σύμβαση του Λουγκάνου του 96 πια. Ε, ή θα πείτε ας προχωρήσει, όποιος προχωρήσει και ένα λόγος θα πάει και η χρηματοδότηση. Κύριε Ονιντή, πολλές ερωτήσεις. Περιμένουμε και τις απαντήσεις σας. Σας ευχαριστώ όλους για αυτές τις ε, πολλές ερωτήσεις. Καταρχήν, τα 70 εκατομμύρια ευρώ που προτείνουμε να δοθούν για αυτό το μέσο χρέους είναι κομμάτι των κονδυλίων που έχουν, που έχουν ψηφιστεί, είναι στο προϋπολογισμό για το 2014, αλλά θα διατεθούν από την 1η Πρώτου ε, του 2015, γιατί τώρα ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με την ε, ε, ΤΕΠ για το σκοπό αυτό. Εδώ όταν μιλάμε για νέο χρηματοδοτικό μέσο, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, δεν βρισκόμαστε σε μια δυναμική όπου πρέπει να επιλέξουμε προγράμματα, αλλά ε, όπου πρέπει να εντοπίσουμε δυνητικά προγράμματα, διότι όπως και εσείς το υπογραμμίσατε, έχουμε πολλά έργα στον τομέα των μεταφορών και προγράμματα τα οποία είναι ενδιαφέροντα για τους επενδυτές γιατί είναι μακροπρόθεσμα και δίνουν ε, ποσοστό απόδοσης ικανοποιητικό. Αλλά δυστυχώς ε, έχουμε και προγράμματα τα οποία είναι εξαιρετικά επικίνδυνα. Και αυτή είναι ακριβώς η φύση των όσων προτείνουμε να τεθεί στη διάθεση των επενδυτών και συμπεριλαμβανομένων των εθνικών αρχών υπάρχει μία διευκόλυνση για να εγγυηθούμε αυτούς τους κινδύνους. Κατά κάποιο τρόπο, και έτσι απαντώ και σε μια άλλη ερώτηση που ετέθη, τα χρήματα αυτά μπορούν να χρησιμεύσουν περισσότερο από ένα προγράμματα με την έννοια ότι τα χρήματα χρησιμοποιούνται μόνο όταν πρέπει να καλυφθεί ο κίνδυνος και όντως δηλαδή ένας επενδυτής δεν μπορεί να έχει τελικά την αναμενόμενη απόδοση από το πρόγραμμα το έργο. Τότε αρχίζει και λειτουργεί η διευκόλυνση αυτή. Και όπως έχετε ζητήσει στη διάρκεια έχετε πει μάλλον στη διάρκεια της συζήτησης, είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε, ε, να προτείνουμε μια τέτοια στήριξη για να μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτού του είδους τα προγράμματα. Ξεκινάμε δηλαδή με κάτι συντηρητικό, προτείνουμε να ξεκινήσουμε με την ΕΤΕΠ που είναι πολύ συντηρητικό παίκτη και με ένα συντηρητικό ποσό επίσης, μόνο και μόνο έτσι ώστε να τροχοδρομηθούν το νέο πρόγραμμα. Αυτό που ελπίζουμε να έχουμε σύντομα και ο Στεφάν εδώ στα δεξιά μου και οι συνάδελφοι συζητάμε εντόνως με διάφορες εθνικές τράπεζες ε, πρόθεσης έργων είναι να είμαστε σε θέση σε συνεργασία με εθνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να δημιουργήσουμε παρόμοια προγράμματα επειδή να βρίσκονται πιο κοντά σε κάποια από τα προγράμματα. Επίσης ρωτήσατε ότι τμήματα αυτών των χρημάτων, στην πρόταση που σας εξήγησε ο κύριο Πρόεδρος Γιούνκερ, τμήμα αυτών των, χρημάτων, δηλαδή 3,3 δις, θα χρησιμοποιηθούν για αυτόν εδώ το σκοπό. Για την ώρα, η Κομισιόν και οι διάφοροι επίτροποι ε, το συζητούν μαζί με τις διάφορες ενδιαφερόμενες επιτροπές, αλλά η ιδέα είναι, για να απαντήσω στην ερώτηση του κ. Ρικέ, είναι να έρθουμε στι αρχές του επόμενου χρόνου με ένα σχέδιο τροποποιητικής νομοθεσίας που θα αποκαλείται Omnibus, γιατί με ένα κείμενο θα τροποποιούνται διάφορα κείμενα, γιατί δεν είναι μόνο ένας κανονισμός, αλλά το και το Horizon 2020, αλλά και το ίδιο το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και γι' αυτό ισχύει η φυσιολογική νομοθετική διαδικασία, οπότε θα έχετε μπόλικο χρόνο να το συζητήσετε μαζί με την Επιτροπή και σε αυτό το χρόνο με το Συμβούλιο. Λυπούμε που δεν μπορώ να πω περισσότερα αυτή τη στιγμή. Η Επίτροπος Μπούλση μάλλον θα θελήσει να αναπτύξει περισσότερο το ε, τις σκέψεις της μαζί σας, ε, ενώπιόν σας. Ε, πάντως θέλουμε αυτό το πρόγραμμα να είναι διαθέσιμο για τον τομέα των μεταφορών και για τα προγράμματα υψηλής προτεραιότητας. Ένα από τα θέματα επίσης ήταν ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτό το μέσο και ένα μέσο equity και αν σκεφτήκαμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε κάποιο τέτοιο μέσο. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα μέσο equity που εξεκολουθεί να έχει μεγάλο δυναμικό και ονομάζεται Marguerite Fund, Ταμείο Μαργαρίτα. Και αυτό θα αναθεωρηθεί εντός δύο ετών, όπου θα εκτιμήσουμε αν θα στηρίξουμε ένα τέτοιο ταμείο για τα προγράμματά μας. Αλλά από την, εκ των προτέρων αξιολόγηση που έχει γίνει και από το είδος των προγραμμάτων που εξετάζει αυτό το ταμείο ε, ημερησίας βάσεως φαίνεται πως το άμεσο ενδιαφέρον είναι ένα μέσο ε, χρεωστικό. Δηλαδή μία διευκόλυνση, μία διευκόλυνση μακροχρόνια. Τώρα, τα διόργες και οι υδατοφράχτες του Άμστερνταμ και σας ευχαριστώ που μου θυμήσατε ότι σήμερα υπάρχει αυτή η παρουσίαση όντως. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Βασίζεται σε χορηγίες για την ώρα το πρόγραμμα αυτό, αλλά ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι τμήμα της στήριξης για αυτό το πάρα πολύ σοβαρό πρόγραμμα και πολύ κρίσιμο πρόγραμμα μπορεί να έρθει και από ένα χρηματοδοτικό μέσο και με πολύ χαμηλότερο κόστος για τις ε, Ολλανδικές Αρχές αλλά και τους διάφορους ε, τέρους στο πρόγραμμα αυτό. Κάθε φορά προσπαθούμε να συζητήσουμε προγράμματα με τα κράτη-μέλη πάντοτε γίνεται μεγάλη προσπάθεια ώστε να πείσουμε τα, τους φορείς να ε, εστιάσουν την προσοχή όχι μόνο στα εύκολα χρήματα που έρχονται με τις επιδοτήσεις αλλά και με το να τους πείσουμε ότι μπορούν να αποφέρουν και όλα αυτά τα προγράμματα. Τα, τώρα μεγάλα προγράμματα όπως το Λιόν, το Ρήνο, το Τούνελ, η σύραγγα του Μπρέναρου κτλ. Ε, το μέγεθος της στήριξης που θα προέρθει από αυτό την διευκόλυνση σε ΕΦ. δεν μπορώ να πω κάτι άλλο παρά το maximum, το, το ανώτατο, η ανώτατη οροφή που προβλέπετε. Βέβαια είναι προγράμματα μεγάλου κινδύνου και που μπορεί να ωφεληθούν όχι μόνο από αυτήν εδώ τη διευκόλυνση, αλλά και από το ε, Ταμείο το ευρύτερο για τις υποδομές που παρουσίασε ο Πρόεδρος Γιούνκερ. Νομίζω πως ε, για όλα αυτά τα προγράμματα υπάρχει δυσκολία βεβαίως τη σήμερα ημέρα να πείσουμε τις εθνικές αρχές να ε, συμφωνήσουν ε, και όλα αυτά είναι υπό το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης δεν αλλάζει κάτι. Το μόνο που προστίθεται υπό την πρωτοβουλία Γιούγκερ είναι μια ρητή αναφορά που προβλέπει εξαίρεση για το ποσό εθνικής χρηματοδότησης που θα επενδυθεί στην στρατηγική διευκόλυνση επενδύσεων. Ένα μικρό άνοιγμα δηλαδή για κάποια ευελιξία στο πλαίσιο του συμφώνου ε, σταθερότητας και ανάπτυξης. Τώρα, αν με αυτό το μέσο θα στηρίξουμε τα προγράμματα που θα ε, υποβληθούν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, όχι. Είναι διαφορετικά. Και πάλι η αίτηση για υποβολή προτάσεων αφορά επιχορηγήσεις και στην φάση της προετοιμασίας των προγραμμάτων προσπαθήσαμε να κατευθύνουμε τους υποψηφίους είτε για τις επιχορηγήσεις είτε για το μέσο χρηματοδότησης. Ξέρουμε ότι θα είναι μεγάλη η συμμετοχή και προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε όσο γίνεται καλύτερα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Αν θα υπάρξει τώρα συγχρονισμός ανάμεσα στην εξπόστα αξιολόγηση που θα γίνει το 2015, εμείς ξεκινάμε αυτήν την εξπόστα αξιολόγηση ήδη τον Ιανουάριο ώστε να γίνουν παράλληλα αυτές οι δύο εργασίες, να μην περιμένουμε δηλαδή μέχρι ότου να εφαρμόσουμε αυτό το νέο, ε, τη νέα χρηματοπιστωτική διευκόλυνση. Γιατί περιμένουμε κάποια προγράμματα να είναι όριμα και να μπορέσουν να υποφεληθούν από τη διευκόλυνση και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και κάποια προγράμματα εκτός των αυτοκινητοδρόμων. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές γιατί τα περισσότερα προγράμματα ήταν ε, για τις οδικές μεταφορές και πιστεύουμε πως έχουμε τη δυνατότητα εδώ και την ευκαιρία να είμαστε τμήμα όλων αυτών και να έχουμε προγράμματα σε πραγματικούς τομείς προτεραιότητας για όλους μας που είναι οι σιδηρόδρομοι αλλά και τα λιμάνια. Βέβαια δεν σημαίνει πως μόνο αυτή η τομή είναι διαθέσιμη για χρηματοδότηση με τη νέα διευκόλυνση. Όχι, γιατί αυτό έχει να κάνει και με την όρεξη των ιδιωτών επενδυτών. Ανέφερα την διευκόλυνση χρηματοδότησης για να μπορέσει να ε, ε, ε, αναπτυχθεί το ERTMS και όντως κύριε Βαντερκάμπ εργαζόμαστε σε αυτήν την διευκόλυνση για να μπορέσουμε να εξυγχρονίσουμε τις μαούνες για τις εσωτερικές πλωτές οδούς. για να αναπτυχθούν δηλαδή και τα συστήματα πληροφορικής ώστε η εσωτερική ναυσιπλοεία να είναι όχι μόνο ασφαλέστερη αλλά και να προσφέρει επιχειρηματικές ευκαιρίες μέσω ενός συστήματος πληροφόρησης που θα είναι διαθέσιμο για όλους τους φορείς του τομέα. Νομίζω πως κάλυψα τα περισσότερα θέματα. Εκτός ίσως κύριε Κράμερ δεν μπορώ να σας πω σήμερα την ακριβή αναλογία των διασυνοριακών προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν υπό το ένα μέσο ή το άλλο. Πάντως μπορώ να σας εγγυηθώ ότι μέσα στην επιλογή των προγραμμάτων στην ανοιχτή υποβολή ε, προτάσεων, στην αξιολόγηση εστιάζουμε την προσοχή στο κατά πόσο αυτά τα διασυνοριακά προγράμματα έχουν άμεσο νόημα όσον αφορά την ολοκλήρωση Τη απαραίτητη επένδυση και από την άλλη πλευρά των συνόρων, γιατί έχετε δίκιο ότι στο παρελθόν έχουμε αντιμετωπίσει διάφορες ε, επενδυτικές ε, προσπάθειες που όμως ε, δεν ολοκληρώθηκαν τα δύο τμήματα όπως έπρεπε και είχαμε διάφορες επιβλαβείς δημιουργώνες μάλλον καθυστερήσεις. Επίση, θα πρέπει στις αρχές του επόμενου χρόνου να γίνει συζήτηση με τους συντονιστέ μας που θα σας παρουσιάσουν ε, το τρίτο πρόγραμμα εργασία για το βασικό δίκτυο. Για κάθε έναν από αυτούς τους διαδρόμους θα γίνει λεπτομερής ανάλυση για το τι χρειάζεται ώστε να εξυγχρονιστούν τα διασυνοριακά προγράμματα και εδώ επίση, στόχος είναι να έχουμε επιπλέον εγγύηση ότι ο χρονισμός της επένδυσης είναι ε, σωστός και από τις δύο πλευρές. Ευχαριστώ. ich... Ε, Ευχαριστώ πολύ και πάλι ο κύριος Ερτού για τις ε, πληροφορίες που μας δώσατε συμπληρωματικά. Μια ακόμη όμως συμπληρωματική ερώτηση και στο συγγνώμη που πρέπει να επανέλθω, αλλά δεν είναι σαφές. Μια επιχείρηση, φύ ή ωμέγα μας λέει αύριο για οποιοδήποτε από τα μεγάλα έργα, Λιόν, Τουρίν, Τωρίνο, Μπρένερ, οτιδήποτε. Θέλω τόσα δις να επενδύσω. Με ποιον τρόπο πρέπει να δράσει αυτός ο ιδιώτης επενδυτής, πρέπει να απευθυνθεί στις εθνικές του αρχές. Και να τους πει Κοιτάξτε, βλέπω ότι είναι ένα τέτοιο έργο κέριο, είναι στο βασικό πυρήνα του δικτύου και εγώ είμαι διτεθειμένος να χρηματοδοτήσω με ιδιωτικά κονδύλια αλλά εφόσον έχουμε είτε από το Μαργαρίτα είτε από το Συνδέοντα την Ευρώπη, ότι με οποιοδήποτε συγκεκριμένο τρόπο εγγυήσει και συμπληρωματικά κεφάλαια. Τι θα γίνει στην πράξη, θα πει το κράτο να ορίστε έχουμε τα ποσά, έχουμε δεσμευθεί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει την προκήρυξή τη σε 6, 8, 10 μήνε του χρόνου. Ε, πρακτικά, πρακτικά, γιατί δεν βλέπω απάντηση. Τι θα γίνει, η διαδικασία ποια θα είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο ιδιώτης επενδυτής που θέλει ενδεχομένω να μπει μέσα σε αυτήν την αγορά. Κύριος Κράμερ. Ο κύριος Ερτού είπε ότι δεν μπόρεσε ο ίδιος να δώσει απάντηση στο ερώτημα. Για να δούμε, ο κύριος Ενιντίν πώς τα καταφέρει. Νομίζω ότι η λογική είναι διαφορετική. Όταν κανείς υποβάλλει μια ε, υποψηφιότητα για να τύχει στήριξης, για να πάρει επιδότηση, συμπληρώνει μια αίτηση, πρέπει να ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής, τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα γιατί υπάρχουν στον κανονισμό. Τώρα, ε, προσπαθεί κανείς να συλλάβει συγκεκριμένα έργα που θα υποφεληθούν από αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα. Για να το κάνει αυτό, ακολουθεί διαφορετική λογική. Τα συντάσσει μαζί με τους ενδυνάμει επενδυτές με βάση τις διάφορες ε, ε, διαθέσιμες διευκολύνσεις. Π.χ. αυτή που προτείνουμε σήμερα, 70 εκατομμύρια δίδονται στο κλάδο των μεταφορών και άρα θα επιτρέψει αυτό την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να έρθει και να βάλει και αυτή συγκεκριμένο ποσό και αυτό το γνωρίζουν οι επενδυτές και υπάρχει ενδιαφέρον γιατί υπάρχει αυξημένη ρευστότητα. Η συζήτηση λοιπόν είναι πια να δούμε ποια έργα ε, προσφέρουν συγκεκριμένη απόδοση σε βάθος χρόνου, κάποιου χρόνου και σε ποιο βαθμό οι εθνικές αρχές οι οποίες ε, είναι και οι κύριες των έργων αυτών είναι έτοιμες να επιτρέψουν σε επενδυτές να έρθουν να συμμετάσχουν είτε με ανάθεση, είτε με παραχώρηση, με συμβίες παραχώρησης, με συγχωρείτε, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, έτσι ώστε να συμμετάσχουν οι ιδιώτες επενδυτές είναι διαφορετική η λογική. Δεν μιλούμε για ε, πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Μιλούμε για το ότι οι επενδυτές γνωρίζουν κάποιες διευκολύνσεις, γνωρίζουν ότι υπάρχουν μέσα διαθέσιμα ε, και αποφασίζουν πώς θα πράξουν. Και έτσι διαμορφώνουν το έργο και χάρη σε τεχνική βοήθεια μπορούμε ε, προς όφελος των εθνικών αρχών να έχουμε καλύτερη προετοιμασία των προτάσεων για τα έργα για να είναι ελκυστικά αυτά στους οικονομικούς επενδυτές. Αυτή την άγουσα ακολουθούμε και είναι κάτι που είναι ενσωματωμένο στην πρακτική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και προφανώς η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα διαπραγματευτεί με τους διαφόρους επενδυτές έτσι ώστε να είναι σωστή η ώρα της οικονομικής εξίσωσης. Ευχαριστώ. Για πολύ σύντομα κυρία Σέντερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα. Έχω δύο ερωτήσεις να θέσω. Η πρώτη έχει να κάνει με αυτό το οποίο διαβάσαμε. Η, όλα αυτά τα κονδύλια του συνδέοντας την Ευρώπη μπαίνουν ε, και συνθλίβονται αν θέλετε μέσα από το πρόγραμμα Juncker. Υπάρχει και το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Όλα αυτά ε, αποτελούν ένα ε, πακέτο που θα εκτινόταν μέσα σε τρία έτη μόνο. Δεν ξέρω αν δεν τα διάβασα σωστά ή δεν τα κατάλαβα καλά, αλλά εμείς μιλούμε για έργα που θα ε, είναι σε βάθος χρόνου, πολύ περισσότερο από ότι τρία χρόνια και μάλιστα έχουν πολύ πιο περίπλοκες συνιστώσεις. Αυτό καταρχάς. Κατά δεύτερο λόγο, ε, αυτή η πρόταση τροποποίηση του προγράμματο εργασιών δεν θα δυσκολέψει την πρόσβαση στα έργα που είχαν ήδη προβλέψει τα κράτη-μέλη. Ήδη είναι πολύ δύσκολη η έβρεση επενδυτών και το να ξεκινήσουν έργα ε, σε εθνικό επίπεδο. Πάντοτε είναι πολύ πιο δύσκολο να πιστεί ένα ιδιώτη επενδύτη, να μπει σε κάποιο δημόσιο έργο και πόσο μάλλον μέχρι σήμερα. Η Επιτροπή παρακαλώ. Η ιδέα η βασική είναι να προσφερθεί ειδική χρηματοδότηση σε διάρκεια τριών ετών. Κάθε έτος περίπου 100 δις θα προβλέπονται για αυτό το νέο μέσον ε, το Ταμείο για Στρατηγικές Επενδύσεις. Το Ταμείο αυτό όμως έχει διάρκεια η οποία θα ξεπεράσει την τριετία. Διότι εάν δεν αξιοποιηθούν τα κονδύλια Και αυτό το λέω γιατί θα πρέπει τα χρήματα αυτά να αξιοποιηθούν για να εγγυηθούν κάποιους κινδύνους από ιδιώτες επενδυτές. Αν λοιπόν δεν χρειαστεί να απορροφηθούν τα χρήματα αυτά ως εγγύησης, θα μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν. Άρα δεν θα διαρκέσει μόνο τρία χρόνια το Ταμείο, αλλά πολύ περισσότερο. Και στην τριετία πάνω ούτως ή άλλως, ανάλογα με την επιτυχία της νέας αυτής πρωτοβουλίας, μπορούμε να την αξιολογήσουμε και να πούμε εάν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της. Κάτι το οποίο σήμερα δεν μπορεί κανείς να δηλώσει. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Θερμά. Έτσι ολοκληρώνεται και αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη και πάμε στο επόμενο που είναι η διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών με στόχο την ασφάλεια των οδικών μεταφορών με εισηγήτρια την κυρία Αιάλα Σέντερ η οποία έχει και το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε ήδη, νομίζω, αναφερθεί στις συνθήκες κατά τις οποίες προέκυψε αυτή η έκθεση είναι νέα έκθεση χωρίς να αναφέρεται σε κάτι το νέο και το καινούριο. Και παρά τις παρατάσεις και το πόσο έχει περιπλακεί όλο αυτό το θέμα, έχουμε καταφέρει να φτάσουμε σε κοινή θέση με το Συμβούλιο. Αυτό είναι δεδομένο και είναι γνωστό. Και τώρα θα πρέπει να αναθεωρηθεί η νομική βάση. Δυστυχώς ευτυχώς. Ε, εν πάση περιπτώσει έχουν γίνει όλα αυτά και φτάνουμε σιγά σιγά ε, στη στιγμή της επίτευξης πολιτικής συμφωνίας χάρη στην πολιτική βούληση της Ιταλικής Προεδρίας αλλά και στην πολιτική βούληση θα έλεγα κυρίως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την οποία θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την ταχύτητά της, για την ταχεία αντίδρασή της. Μέσα σε λίγους μήνες κατάφερε να μας παρουσιάσει ένα κείμενο που να ακολουθεί τις γραμμές και τις προτάσεις του δικαστηρίου χωρίς να κάνει το περιεχόμενο πολύ πιο ε, περίπλοκο. Από εκεί και πέρα, η Ιταλική Προεδρία προσπάθησε να υπάρχει συμφωνία στο Συμβούλιο, να μην περιπλακεί περισσότερο το θέμα και να προσαρμοστούμε όλοι στα, στις επιταγές του δικαστηρίου. Και έτσι ε, θα καταφέρουμε ενδεχομένω να τροποποιήσουμε το κείμενο να έχουμε μεγαλύτερη συνειδητοποίηση του τι διακυβεύεται και θα είμαστε σε θέση να ε, αποφύγουμε επιτέλους αυτή την ατιμορρησία των οδηγών που είναι κάτοικοι σε μία χώρα μέλος και διαπράττουν οδικές παραβάσεις σε άλλη χώρα μέλος και τελικά δεν μπορούν να βρεθούν ποτέ. Από εκεί και πέρα θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους που διάβασαν το κείμενο που υπέβαλαν προτάσεις τροποποίησης του και θέλω να πω καταρχάς ότι ορισμένες από τις τροπολογίες αυτές δυστυχώς δεν μπορώ να τις λάβω υπόψη. Ε, τις τροπολογίες της κυρίας Αχνότου γιατί προσπαθεί να επανεθνικοποιήσει κάπως το θέμα και το κατανοώ με δεδομένο την πολιτική ομάδα στην οποία ανήκει, ωστόσο είναι ευρωπαϊκή η οδηγία με την οποία καλούμαστε να ασχοληθούμε και από εκεί και πέρα προσπαθεί να διαγραφούν ορισμένες βασικές έννοιες από το κείμενο. Βασικές έννοιες που έχουν να κάνουν με την οδική ασφάλεια, όπως για παράδειγμα ο οδηγός όταν χρησιμοποιεί το κινητό του τηλέφωνο όταν οδηγεί, όταν μπαίνει σε ε, δρόμο όπου απαγορεύεται η διέλευση και όπου η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας ξεπερνάει τα 50 χιλιόμετρα. Αυτά είναι βασικές έννοιες και δεν μπορώ να, τα, να δεχθώ να μην υπάρχουν στο κείμενο. Μιλούμε επίσης, γίνεται λόγος και για τις ενώσεις ή Συλλόγου συλλόγου των αυτοκινητιστών ή εποχούμενων. Γίνεται αναφορά σε όλους τους παράγοντες, ωστόσο εμείς είχαμε ρητός αναφερθεί στους συλλόγους που ασχολούνται με τα θύματα του αυτοκινητόδρομου. Ε, νομίζω ότι είναι μια διατύπωση η οποία είναι πολύ πιο ακριβής και ταιριάζει περισσότερο στο κείμενο. Επομένως δεν θα δεχθώ αναφορά σε συλλόγους γενικώς αυτοκινηστικών παρά μόνο σε συλλόγους που έχουν να κάνουν με τα θύματα και τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Από εκεί και πέρα έχουμε και την εμπειρία του επαγγελματία οδηγού. Αυτά είναι γνωστά όμως δεν είναι εδώ το κατάλληλο κείμενο για να καλυφθεί το θέμα των πλαστών αδειών οδήγησης. Μιλούμε για τις θεμελιώδεις και βασικές αρχές, στις οποίες οφείλεται το 90% των αυτοκινηστικών ατυχημάτων ή δυστυχημάτων όπου έχουμε θύματα ή τραυματίες. Ε, το θέμα των πλαστών αδειών οδήγησης θα πρέπει να λυθεί ε, σε άλλο νομοθετικό κείμενο. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Φώστερ έχουμε την πρόταση του Συμβουλίου σε σχέση με τις τρεις νέες χώρες που, κάνουν opt-in, που διαλέγουν επιτέλους να εφαρμόσουν αυτή την οδηγία με την καινούρια νομική βάση, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία και η Δανία. Αυτό είναι καλό, ωστόσο νομίζω ότι με την πρότασή μου ε, έχοντας μιλήσει και με όλου τους ενδιαφερόμενους φορείς, καλύπτουμε καλύτερα το θέμα, έτσι όπως είναι διατύπωση του κειμένου αυτή τη στιγμή. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω και δεν επιθυμώ να επιμείνω να πρέπει να περιμένουν δύο χρόνια. Σίγουρα υπάρχουν συμφέροντα που θέλουν να καθυστερήσουν τη θέση σε ισχύ ε, της οδηγίας, της νέας οδηγίας και έχουμε και την αναθεώρηση του 2016. Έχω πάρα πολλές επιφυλάξεις λοιπόν και προτιμώ τη δική μου διατύπωση. Ε, την διατύπωση που ε, στην οποία έχουμε καταλήξει η κυρία Άντερσον και εγώ. Δηλαδή ένας χρόνος να είναι το μεταβατικό χρονικό διάστημα μέχρι ότου να μπορέσουν αυτές οι τρεις χώρες να την υιοθετήσουν και να τη θέσουν σε ισχύ και όχι δύο χρόνια. Νομίζω ότι οι τρεις αυτές χώρες μπορούν να κάνουν περισσότερα για να ε, δυναμώσουν την οδική ασφάλεια. Ήδη το κάνουν, δεν θα πρέπει να είναι τεράστιο πρόβλημα να ενσωματώσουν την οδηγία μέσα σε ένα χρόνο στο δικό τους δίκαιο. και η έκθεση αναθεώρησης μάλλον θα πρέπει να ε, παραταθεί από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή θα είναι η πρότασή μου σε γενικές γραμμές. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, Ζόρς Μπαχ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και νομίζω ότι μπορώ να συμφωνήσω με τα όσα είπε η κυρία Γιάλα Σέντερ Πιστεύω ότι ιδιαίτερα ευχόμαστε όλοι οι εμπλεκόμενοι να προχωρήσει γρήγορα η υπόθεση αυτή για την ασφάλεια των οδικών μεταφορών. Συμφωνώ με τις ε, απόψεις που εξέφρασε η ΝΕΣ ε, για τις τροπολογίες. Το, ε, η προσπάθεια για την επανεθνικοποίηση θα ήταν αντιπαραγωγική εν προκειμένου και οι κύριες πτυχές της ασφάλειας των οδικών μεταφορών θα πρέπει να ε, αναφέρονται ξεκάθαρα και αυτό αναμφίβολα για μένα. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα λοιπόν, ε, όπως άλλωστε επεσήμανε και η, ε, η συγγήτρια, θέλει με την ε, τροπολογία 17 να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Πέτερ Φαντάλεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι καιρός να ολοκληρώσουμε με αυτό το θέμα που έχουμε τόσο καιρό στην ημερησία μας διάταξη. Είναι απαραίτητο όχι μόνο προς το συμφέρον της οδικής ασφάλειας, αλλά και διότι αν υπάρχουν παραβάσεις, οι ε, οδηγοί θα πρέπει να ε, είναι υπόλογοι για αυτές. Συμφωνώ λοιπόν με τον εισηγητή ότι θα πρέπει να προσέχουμε να μην ξανανοίξουμε ολόκληρη τη συζήτηση και να την επαναλάβουμε πράγμα για το οποίο διστάζει για τις διάφορες τροπολογίες ε, συμφωνώ με την ε, δισταγμούς αυτούς και εγώ αλλά ξέρω ότι η κυρία Φώστερ θα ήθελε να έχουμε περισσότερο χρόνο στην ομάδα μας πάντοτε ε, συζητάμε το θέμα αυτό. Εγώ είμαι έτοιμος για κάποια μεγαλύτερη ευελιξία, αλλά ε, συμφωνώ ότι δεν πρέπει να επανέλθουμε στην αρχή, στην αφετηρία, με όλες αυτές τις τροπολογίες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Κούν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Για να καταλήξει η ομάδα μας σε συγκεκριμένη θέση θα πρέπει να σας πω ότι θα ε, έχουμε συνοχή σε σχέση με αυτά που έχουμε πει εξ αρχής. Πρέπει να εφαρμόσουμε την απόφαση του δικαστηρίου. Συμφωνώ με την εισηγήτρια, με τη συντάκτρια της ε, έκθεσης αυτής. Στη δική μου πολιτική ομάδα ανέλαβα τη δέσμευση να μην υποβάλλουμε καθόλου τροπολογίες, γιατί το επίγον είναι να εγκριθεί η έκθεση ως έχει και στη συνέχεια να έχουμε σύνταξη έκθεσης για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκε η νέα οδηγία το 2006 και σε αυτή την καινούργια έκθεση τότε το 2006 να κάνουμε την κριτική μας. Θεωρώ λοιπόν ότι ορισμένες χώρες υιοθετούν τους, ε, τους κανονιστικές αυτές διατάξεις, υπάρχει νομική ανασφάλεια, εμείς θα απορρίψουμε όλες τις τροπολογίες και θα υπερψηφίσουμε μόνο ε, τροπολογίες που προβλέπουν όσο το δυνατόν πιο ε, ασφικτικές και στενές προθεσμίες. Και γι' αυτό προτιμούμε να έχουν αυτές οι τρεις χώρες που επιλέγουν να ενσωματώσουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο ένα χρόνο προθεσμία να το κάνουν και όχι δύο. Από εκεί και πέρα συμφωνώ απολύτως με την εισηγήτρια και το έχω δείξει σε όλες τις συναντήσεις που είχαμε μεταξύ μας. Ευχαριστώ. Η κυρία Καρίμα Εντέλη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, την εισηγήτρια. Ε, εξ ονόματος των οικολόγων θα ήθελα να πω ότι η πρόταση που υποβάλλεται είναι καλή. Εμείς συμφωνούμε Ωστόσο, σας υπενθυμίζω ότι έχουμε χάσει πάρα πολύ χρόνο. Ε, έχει έρθει πλέον η ώρα να υιοθετήσουμε, να εφαρμόσουμε την νομοθεσία. Συμφωνώ μαζί σας ε, σε όλες αυτές τις βελτιώσεις που θέλετε να επιφέρετε ε, σε, σε συμφωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτό ευχαριστώ. Και η Μαρή Κριστίνα Αρνότου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια διότι υπογραμμίζει ε, ότι είχα στο μυαλό μου πράγματι τους Γάλλους αυτοκινητιστές ε, καταρχάς και όντως μπορεί αυτό να συμβαίνει, ωστόσο εσείς γελιοποιήσατε τις τροπολογίες μου και θα προσπαθήσω να ε, τις εξηγήσω. Είναι 12 οι τροπολογίες. Συμφωνούμε και θέλουμε τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για την οδική ασφάλεια. Ωστόσο, δεν είναι καθήκον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προβλέπει ε, κανονισμούς απομόνητες, είτε μιλούμε για τα ραντάρ, είτε για ε, την πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων ε, ε, σε περιπτώσεις διάπραξης παραβάσεων και ούτω καθεξής. Μπορεί αυτό να τα κάνουν τα κράτη-μέλη πάρα πολύ καλά από μόνα τους και η αρχή της επικουρικότητας δυστυχώς εδώ καταστρατηγείται. Σύμφωνα με το κείμενο, οποιαδήποτε πολιτική ε, οδική πρέπει να, είναι, να, περιβα... επιβάλλει μεγαλύτερους περιορισμούς. Αυτή, είναι, η ιδεολογική προσέγγιση. Ε, δεν είναι πολιτική. Το μόνο που κάνει είναι να μην λαμβάνει υπόψη της τις τοπικές ιδιωτερότητες και να γονατίζει όσους ε, χρησιμοποιούν οχήματα για τη μεταφορά τους. Και βεβαίως θα πρέπει να προβλέπεται ο σωστός προϋπολογισμός για τους ε, οδούς ε, και αυτή την κατάσταση τη βιώνουμε στη Γαλλία κάθε φορά που έρχεται ο χειμώνας, κάθε χρόνο. Θα πρέπει λοιπόν οι εκπρόσωποι όλων αυτών που ασχολούνται με το αυτοκίνητο να ε, συμμετέχουν στη συζήτηση και να του ζητείτε η γνώμη ε, σε ισότιμη βάση. Δεν μίλησα για, τις, ε, για την υπέρβαση του όριου ταχύτητας πέραν των 50 χιλιόμετρων. Είπα αντίθετα ότι όταν κάποιος ξεπερνάει το όριο ταχύτητας μόνο κατά 5 χιλιόμετρα, ε, δεν θα πρέπει να του επιφυλάσσουμε την ίδια μεταχείριση με αυτή που έχουμε για κάποιον που ε, ξεπερνάει το όριο ταχύτητας κατά 50 και χιλιόμετρα. Άλλο οι μικρές παραβάσεις και άλλο η ουσιαστικά η εγκληματικότητα, όπως το Go Fast που είναι μέθοδος που χρησιμοποιούν οι έμποροι ναρκωτικών για να μεταφέρουν τα ναρκωτικά τους. Δηλαδή, ε, ε, πηγαίνουν από το ένα σημείο στο άλλο με δύο οχήματα, ε, πολύ μεγάλης υποδύναμης. Το ένα μεταφέρει τα ναρκωτικά και το άλλο όχι. Είναι λοιπόν παραβατικότητα μεγάλη εδώ, εγκληματικότητα, δεν έχει σχέση μόνο με την ε, παράβαση του ΚΟΚ και θα πρέπει όλα αυτά να τα τονίσουμε. Να έχουμε περισσότερη ευελιξία με τους ε, κανονικούς εποχούμενους και μεγαλύτερη αυστηρότητα έναντι των εγκληματιών και των παραναβατών. Αυτό ήταν το νόημα των τροπολογιών μου. Ευχαριστώ. Λούση Ευχαριστώ, άκουσα με χαρά το ότι προβάλλει αυτή την οδηγία για το χρονικό περιθώριο για τα τρία κράτη-μέλη συγγετρία, αυτά που δεν είχαν αρχικά προβλεφθεί. Βέβαια, αντιλαμβάνομαι ότι θα υπάρχουν κάποιε προποθέσει τεχνικέ διοικητικέ, οι οποίε θα πρέπει να συμμορφωθούν. τι κοιτάω στι λεπτομερίε τους, ανησυχίε που έχουν να κάνουν με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ενώ υπάρχουν κάποιε άλλε ρυθμίσει. Ε, που καλύπτουν πιστεύω τις ανησυχίες. Υπάρχει ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την εξασφάλιση της ε, υποδομής της ε, μηχανογράφησης, της πληροφορικής. Αυτό νομίζω ότι μέσα σε ένα χρόνο αντί για δύο μπορούν να το καταφέρουν και νομίζω ότι είναι λογική η προσέγγιση δεδομένου δε ότι η αξιολόγηση δείχνει ότι μπορεί να έχει κρίσιμη σημασία και να σώσει πολλές ζωές στην Ευρώπη αυτή η οδηγία, η εφαρμογή της. Συμφωνώ λοιπόν με εκείνους οι οποίοι λένε ότι θα πρέπει να είναι ώστε να τον πιο μικρές οι καθυστερήσεις. Γι' αυτό λοιπόν χαίρομαι ιδιαίτερως και πρέπει να πω ότι υπάρχει μια τροπολογία για την παράνομη χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλων μέσων ε, επικοινωνίας Κάποιοι συνάδελφοι φαίνεται να έχουν διαγράψει, δηλαδή δεν θέλουν να υποστηρίξουν την ασφάλεια. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να επιμείνουμε και να επανέλθει το μέτρο αυτό και να υποστηριχθεί η τροπολογία 17. Ευχαριστώ, Φώστερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον, την εισηγητρία. Θέλω να επαναλάβω το εξής. Στην προηγούμενη συνεδρία με την ανταλλαγή απόψεων είχατε τυπώσει μια αίτηση σχέση με την εφαρμογή και το χρονικό περιθώριο που θα δοθεί στα τρία κράτη που δεν είχαν αρχικά καλυφθεί από το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία. Όλα τα κράτη είχαν δύο χρόνια προσαρμογή. Όμω το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία και η Δανία αφού συμφώνησαν πλέον και θα συμπεριληφθούν, θα σταματήσει η παρέκκληση δηλαδή, δεν θα υπήρχε η παρέκκληση αυτά, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν πρέπει να έχουν τα δύο χρόνια που είχαν και οι άλλοι δύο ως χρόνο προσαρμογής. Και αυτό σας το λέω όχι γιατί κάποιος προσπαθεί ε, επαόριστο να αναβάλει την εφαρμογή του συστήματος, αλλά γιατί στο Ρωμένο Βασίλειο θα χρειαστεί πρωτογενές δίκαιο, λέει η ομιλήτρια, για να προσαρμοστούμε και να εφαρμοστεί η οδηγία. Γιατί και η Γερμανία, ξέρετε, έχει αντίστοιχα αντίστοιχη νομοθεσία. Χρειάστηκε τα δύο χρόνια για να κάνει σωστά την προσαρμογή της. Και άρα η τροπολογία που πρέπει να πω, κυρία Ιασάντερ, δεν το περίμενα αυτό. Δεν βλέπω και για ποιο λόγο. Αν χρειαστούν κάτι παραπάνω από ένα χρόνο τα κράτη-μέλη, αν πάνω στους 18 μήνες πειράζει, μπορεί να είναι και λιγότερο από δύο χρόνια. Τόσο το καλύτερο. Εάν όμως ισχύσει μήνο ή αλλιώς την πατήσατε, τι θα τους κάνουμε δηλαδή αν δεν μεταφέρουν τις ε, διατάξεις μέσα σε ένα 12 μήνο, θα τους επιβάλλουμε κυρώσεις, θα τους τιμωρήσουμε. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν δυσκολίες. Ο καθένας έχει την ένωμη του τάξη, το νομικό του σύστημα. Δεν έχει κανείς ε, πιο πολύ δίκαιο από τον άλλον ή κάποιος λιγότερο. Πρέπει να αρχίσουμε να συμπεριφερόμαστε σαν όριμοι και ενήλικες άνθρωποι και να κοιτάξουμε να κάνουμε τη δουλειά μας στα σοβαρά. Δεν θέλει κανείς να μην βελτιωθεί η οδική ασφάλεια. Εμείς έχουμε άλλωστε στον Ηνωμένο Βασίλειο πολύ καλές επιδόσεις. Αλλά μην ξεχνάμε δεν είναι μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία και η Δανία επίσης. Και για τους λόγους που σας εξήγησα πρέπει να έχουν περισσότερο χρονικό περιθώριο. Ευχαριστώ την εισηγήτρια βεβαίω και ελπίζω να λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις μου. Σας ευχαριστώ. Τσίντσκα. Digimove. Yes, uh, thank you, Mr. Chairman. Good, good... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και ολόκληρη την Επιτροπή Μεταφορών για την εξαιρετική εργασία που έχετε κάνει σε αυτό το σχέδιο οδηγίας. Θα ήθελα να θυμίσω αυτά που είπα σε προηγούμενη συνεδρίαση όταν παρουσιάστηκε η έκθεση, ότι πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου προσπάθεια στην οποία κατέληξαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο. Εμείς έχουμε μεγάλη στήριξη ε, βεβαίω ε, ανέκαθεν για το σημαντικό θέμα της οδικής ασφάλειας. Όταν ε, η Κομισιόν λοιπόν ε, έκανε το σχέδιο πρότασης μετά από την απόφαση του, του δικαστηρίου της 6ης Μαΐου, στόχος ήταν να εξασφαλίσουμε ότι μέχρι τις 6 Μαΐου 2015 δεν θα υπήρχε πλέον νομικό κενό στην Ευρώπη όσον αφορά την διασυνοριακή επιβολή των προστήμων. Ε, Τώρα έχουμε μια πολύ καλή έκθεση της ηγήτριας και εμεί εξασφαλίσαμε και ένα καλό πρόγραμμα από το Συμβούλιο αρχές Οκτωβρίου. Όσον αφορά τις τροπολογίες που υπευλήθησαν, η Κομισιόν είναι εξαιρετικά ικανοποιημένη με την τροπολογία 1, διότι πιστεύουμε πως η τροπολογία αυτή διορθώνει την γνωμοδότηση EDPS και ταιριάζει στο ευρύτερο πλαίσιο που αφορά την προστασία των δεδομένων. Μπορούμε να δεχτούμε την τροπολογία 2 που πιστεύουμε είναι μια μικρή τεχνική ε, τροπολογία. Όσον αφορά τις δύο τροπολογίες τώρα που αφορούν την ε, το χρόνο μεταγραφής που επιτρέπουν ε, περισσότερο χρόνο στα κρατημέλη για τη μεταγραφή της οδηγίας. Η Κομισιόν είναι φυσικά έτοιμη να δεχτεί κάποια ευελιξία σε σχέση με αυτά τα τρία κρατημέλη, διότι διαπιστώνουμε ότι θα χρειαστούν λίγο περισσότερο χρόνο για την ε, μεταγραφή της. Και για τις υπόλοιπες τροπολογίες θεωρούμε, έχουμε εξετάσει πολύ προσεκτικά τις έχουμε εξετάσει πολύ προσεκτικά, αλλά κατά τη γνώμη μας ξεπερνούν την αρχική αντίληψη για αυτό το συγκεκριμένο σχέδιο οδηγία. Δεν θέλαμε εμείς να ξεπεράσουμε το αρχικό κείμενο, στόχο είχαμε μόνο να διορθώσουμε την νομική βάση και έτσι θα θέλαμε να ζητήσουμε από την Επιτροπή να μην στηρίξει αυτές τις άλλες τροπολογίες. Εάν μπορώ να πω ακόμα κάτι στο τέλος, θεωρώντας ότι αύριο θα υπερψηφιστεί η πρόταση, θα γίνει τριμερής διάλογος στις 11 Δεκεμβρίου. Και ελπίζουμε πραγματικά ότι αυτό ο τριμερής θα είναι επιτυχής και θα επιτευχθεί συμφωνία ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο. Και ακόμα και αν είμαστε μόνο Δεκέμβριο, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε από πλευρά των τριών θεσμικών οργάνων ότι θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία σου γίνεται πιο σύντομα, διότι θα ήθελα να σας θυμίσω ότι στις 6 Μαΐου του επόμενου έτους δεν θα υπάρχει πια νομική βάση για την ε, επιβολή, τη διασυνοριακή των ε, προστήμων κυκλοφορίας. Θα ήθελα λοιπόν αυτό να σας το θυμίσω οργανωτικά έτσι ώστε στην διοργάνωση των επόμενων στάδιων της ψηφοφορίας, εάν θεωρήσουμε βέβαια ότι ο τριμερής θα είναι θετικός, να πάμε στην Ολομέλεια όσο γίνεται πιο γρήγορα, ώστε να μην υπάρξει καθυστέρηση και να μην βρεθούμε άνευ νομικής βάσης μέχρι τις 6 Μαΐου. Ολοκληρώνω ευχαριστώντας ακόμα μια φορά τον εισηγητή και όλα τα μέλη της Επιτροπής Μεταφορών για την εξαιρετική σας δουλειά. Ευχαριστώ η κυρία Σέντερ, Αγιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ και εγώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τα σχόλιά σας και θέλω να κάνω δύο διευκρινήσεις. Πρώτον, σε σχέση με τα σχόλια της κυρίας Φώστερ, να σας υπενθυμίσω ότι από το 2007 τρία χρόνια περιμέναμε, γιατί ορισμένες κυβερνήσεις πράγματι δεν ήθελαν αυτή την οδηγία. Και η νομική βάση της οδηγίας ήταν οι μεταφορές ακριβώς για να μπορεί να προχωρήσει. Και τελικά η Βελγική Προεδρία είχε την καταπληκτική ιδέα να αλλάξει η νομική βάση της οδηγίας και έτσι να μπορέσει να προχωρήσει η οδηγία αυτή. Εκτός ε, των τριών χωρών που είχαν προβλήματα. Προχωρήσαμε. Μετά το δικαστήριο ε, θεώρησε ότι οι τρεις αυτές χώρες που είχαν κάνει opt-out πρέπει να μπουν και να την εφαρμόσουν λόγω της διαφορετικής νομικής βάσης. Επομένως δεν είναι αφελές ούτε παιδαριώδες αυτό που λέω, απλά δεν έχω εμπιστοσύνη πλέον και το καταλαβαίνετε αυτό, ε, ότι πιστεύω ότι δεν χρειάζονται δύο χρόνια οι χώρες αυτές ή τόσο προηγμένες, μπορούν μέσα σε ένα χρόνο να το ενσωματώσουν ε, στην εθνική τους νομοθεσία, ειδικά το Ηνωμένο Βασίλειο. Και επειδή δεν έχω πια εμπιστοσύνη σε κανέναν, θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε ε, πολύ αυστερά ε, μέτρα έτσι ώστε στο προσεχή τριμερή διάλογο το Συμβούλιο να μην βγάλει κι άλλο άσο από το μανίκι του αν θέλετε. Και γι' αυτό ελπίζω οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου ε, να μην χρειαστεί να αντιμετωπίσουν ε, τέτοιου είδους καταστάσεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό θα φανεί. Στην κυρία Αγνό του ε, λέω ο, ε, το εξή. Ποτέ δεν έχω γελιοποιήσει καμία τροπολογία από κανένα συνάδελφο, από καμία πολιτική ομάδα και εσεί θα πρέπει να ε, σκεφτείτε και να προβληματιστείτε για το πώς αναγνωρίζετε αυτούς που οδηγούν οχήματα και δημιουργούν πολύ σοβαρά προβλήματα στην οδική ασφάλεια από τη μία και από την άλλη το όραμα που έχουμε για να μειώσουμε ε, τους, ε, τα χιλιάδες θύματα που πληρώνουν το φόρο της ασφάλτου. Οι λαθρέμποροι ναρκωτικών δεν, οφείλονται ε, δεν ευθύνονται αυτοί για αυτά τα χιλιάδες θύματα που έχουμε κάθε χρόνο στην Ευρώπη. Σαφώς και πρέπει να τιμωρούνται, αλλά δεν είναι αυτό το βασικό θέμα από πλευράς οδικής ασφάλειας. Θα πρέπει όλοι να εκπροσωπούνται πράγματι και οργανώσεις αυτοκινηστιών ή εποχούμενων και ε, το σημαντικότερο κατά τη γνώμη μου είναι ε, να ακούσουμε τη φωνή αυτών που έχουν υποφέρει περισσότερο και που αγωνίζονται καθημερινά για να βελτιώσουν την ασφάλεια στους δρόμους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έτσι ολοκληρώνεται αυτό το σημείο στην ημερησία μας διάταξη. Αύριο προβλέπεται η ψηφοφορία. Να είσαστε όλοι παρόντες, ελπίζω. Τώρα βλέπω ότι από το ΕΛΚ μπορεί να είναι περισσευούμενος, αυτό το ρυθμίσουμε αύριο. Τώρα έχουμε λοιπόν την παρουσίαση του, της ηλεκτρονικής συνεδρίασης, e-meeting από την DG έχετε το λόγο και έχει πολύ χαιρόμαστε που σας βλέπουμε και εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα κάνω μια σύντομη παρουσία σας για ένα νέο εργαλείο που θα σας βοηθήσει στη δουλειά σας εδώ στην ε, ε, Επιτροπή. Το όνομά του είναι e-meeting, ηλεκτρονική συνεδρίαση. Είναι τμήμα της εργασίας άνευ εγγράφων, χαρτιού δηλαδή. Η παρουσίαση θα είναι πολύ πολύ σύντομη και καλώ όλους με το κινητό κινητή του συσκευή να με ακολουθήσουν. Πρόκειται για μια εφαρμογή που βασίζεται στο δίκτυο και λειτουργεί σε οποιαδήποτε συσκευή και επίσης είναι προσβάσιμο σε οποιαδήποτε στιγμή. Θα σας δείξω αμέσως ε, το διαφημιστικό, το demo. Θα σας δείξω το... Πρέπει να μπούμε στο site του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθετος ή e-meeting. The Η ίδια η εφαρμογή είναι εσωτερική, δηλαδή είναι προσιτή μόνο στο προσωπικό ε, του Κοινοβουλίου, στους Ευρωβουλευτές και στους βοηθούσες. Έχουμε λοιπόν εδώ τους διάφορους κωδικούς, το όνομα χρήστη, Μπορείτε όλοι να δείτε και το δικό μου κωδικό τώρα. Πρώτη φορά όταν έχετε πρόσβαση λοιπόν στην εφαρμογή βλέπετε αυτή την οθόνη. Είναι μια εισαγωγική οθόνη που λέει ότι είναι τρία τα βήματα για να έρχεται πρόσβαση στα έγγραφα. Ξεκινώ λοιπόν πιέζοντας το start. Ε, στα πάνω αριστερά στη σελίδα έχουμε μια ειδοποίηση για τις γλώσσες, γιατί υπάρχει σε όλες τις γλώσσες είναι διαθέσιμη αυτή η εφαρμογή. Δίπλα εκεί Επίσης λέει ότι είναι διαθέσιμο για όλες τις επιτροπές. Σήμερα ας πούμε πάω στην Επιτροπή Μεταφορών Ορίστε. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε επιλέξει την Επιτροπή Μεταφορών θα πάει το σύστημα στον μήνα, στον τρέχοντα μήνα και ε, αναφέρει όλες τις ε, συνεδριάσεις που προβλέπονται και στα αριστερά την ημερήσια διάταξη. Ε, την, ε, τα κείμενα που υπάρχουν, δηλαδή η μερίσια διάταξη. Έχουμε, αν θέλουμε, αν, βάλουμε, αν χτυπήσουμε το συν, έχουμε έξτρα πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα που θα εξεταστεί και βέβαια το όνομα του εισηγητή, του σκιώδους εισηγητή και ούτω καθεξής. Εδώ λοιπόν μπορούμε να δούμε την ημερήσια διάταξη σε πλουσιότερη μορφή. Μπορούμε επίσης να περάσουμε στην εικόνα, να δούμε μάλλον τα έγγραφα. Εκεί βλέπουμε τα έγγραφα μόνο, δεν έχουμε πια πληροφορίες επιπλέον για την ατζέντα. Και πάλι εδώ έχουμε ένα ευρετήριο, ένα ευρετήριο που φανταστείτε ας πούμε στη διάρκεια μιας συνεδρίσης θέλει κανείς να προσαρτήσει ένα έγγραφο για να συζητηθεί, να το παρουσιάσει μάλλον για να συζητηθεί. Δεν χρειάζεται πια να αγχωθούμε. Πρέπει, μπορεί η γραμματεία αμέσως να ανεβάσει το έγγραφο και να έχουν όλη πρόσβαση σε αυτό. Αυτό λοιπόν είναι ένα ωραίο τρόπο να έχουμε σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα έγγραφα. Το e-committee, η ηλεκτρονική συνεδρίαση μπορεί να, είναι ένα, να δώσει πρόσβαση μάλλον και στο μεγαλύτερο, ευρύτερο intranet της Επιτροπής Μεταφορών όπου μπορεί κανείς να αναζητήσει όλα τα έγγραφα. Αλλά εστιάσουμε τώρα στο e-meeting. Έχουμε και άλλο ένα, μια δυνατότητα. Μπορούμε δηλαδή να μοιραστούμε τα σημεία της ημερήσιας διάταξης. Για παράδειγμα, λέει εκεί η συνεδρία συντονιστών, κάνω κλικ εκεί και το σύστημα μου επιτρέπει να το μοιραστώ. Μαζί σας. Τώρα δεν λειτουργεί, αλλά κανονικά λειτουργεί. Επανέρχομαι λοιπόν στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Όλα τα έγγραφα εδώ είναι προσιτά σε διάφορες γλώσσες. Για παράδειγμα, εδώ έχουμε τις τροπολογίες και η εφαρμογή αυτή είναι διαθέσιμη πριν αλλά και μετά τη συνεδρίαση. Δηλαδή μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση σε συνεδρίαση της περασμένης χρονιάς ή πριν τη συνεδρίαση να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε γλωσσική εκδοχή που έχει μεταφραστεί. Παράδειγμα, ανοίγω αυτό εδώ το έγγραφο σε οποιαδήποτε γλώσσα το σύστημα ανοίγει το έγγραφο προς ανάγνωση. Εδώ λοιπόν η εφαρμογή σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στο έγγραφο. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε περισσότερο με το συγκεκριμένο έγγραφο, μπορούμε να το ανοίξουμε σε μια άλλη εφαρμογή. Για παράδειγμα, μπορώ να το ανοίξω σε αυτή την εφαρμογή που έχω εγώ στη δική μου συσκευή και μετά μπορώ να προσπαθήσω να το επεξεργαστώ. Σαν να ήταν χάρτινο το έγγραφο μπορώ να σημειώσω επάνω του, να διορθώσω, να αλλάξω και να προσθέσω και το σχολείο μου. Εδώ λοιπόν είναι ο τρόπος με τον οποίο εργαζόμαστε πάνω στα έγγραφα. Όταν έχω κλείσει, τελειώσει, μπορώ να το μοιραστώ με το βυθό μου, του συναδέλφους μου και όλα τα έγγραφα που έχω, μάλλον όλα τα σχόλια και οι σημειώσεις που έχω κάνει πάνω στο έγγραφο παραμένουν σε αυτόν τον φάκελο που είναι προσδεδεμένος, το έχω κάνει attachment και μπορώ να το μοιραστώ με όλους σας. Και τα σχόλιά μου είναι ιδιωτικά. Κανείς άλλος δεν θα δει τι αλλαγέ εκτός γιατί έχω κατεβάσει το κείμενο στη συσκευή μου, σε άλλη εφαρμογή, σε άλλο application και κανείς δεν μπορεί να δει τα σχόλιά μου, εκτός από αυτούς που εγώ θέλω να τα στείλω. Αν νόμιζα είχε ερώτηση. Όχι. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα Χαρακτηριστικό σενάριο για πρόσβασης λοιπόν στα έγγραφα της συνεδρίασης και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ θέλω να συγχαρώ την ε, DG Tech, γιατί από τότε που έφτασα εδώ έχω εντυπωσιαστεί απίστευτα με τις υπηρεσίες σας, τις ε, ικανότητες, ε, την ε, υπηρεσία που προσφέρετε στο μέλη, ε, που βελτιώνεστε και, βοηθάτε, είστε όλοι πολύ ευγενικά, έχετε πρόσβαση σε διάφορες μορφές ε, pads και ταμπλέτας και αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι πώς αυτό συνδέεται με το νέο σύστημα διαχείρισης της γνώσης που αναπτύσσεται και ενθαρρύνεται και επίσης χρειάζεστε, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλα αυτά μέσω κάποιο πόρταλ στο βασικό browser ή χρειάζεται κάποιο token ή κάποια ειδική πρόσβαση για να μπει κανείς σε αυτό το σύστημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Καταρχήν, η εφαρμογή είναι εσωτερική για την ώρα. Δηλαδή, θεωρείται εσωτερικός πόρος. Για να έχουμε πρόσβαση σε αυτήν έχουμε δύο τρόπους. Είτε μέσω των τερματικών που έχουμε, σαν να ήταν ε, desktop, είτε μέσω του δικού μας πόρταλ ε, του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι ένα είδος extranet. Εδώ βασιζόμαστε στο, στο όνομα και στο κωδικό, αλλά θα ενισχύσουμε την ασφάλεια για να ε, προσθέσουμε άλλο ένα στρώμα, άλλο ένα επίπεδο ασφάλειας. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή ε, προσπαθούμε να καταστήσουμε την πρόσβαση σε όλα αυτά τα συστήματα όσο γίνεται πιο εύκολα. Τώρα, επειδή είμαστε στη πιο τη φάση της ε, παροχής όλων αυτών των ε, ταμπλετών, όταν γράφεται μια συσκευή υπάρχει ένα είδος εμπιστοσύνης και αυτό επιτρέπει και την πρόσβαση. Τώρα για τη διαχείριση της γνώσης στο άλλο πρόγραμμα ένα μεγάλο κομμάτι αυτού έχει να κάνει με συνεργασία για τις πολιτικές ομάδες και για τις επιτροπές, γιατί θα είναι αυτός ο χώρος όπου κανείς πρέπει να προετοιμάσει όλα αυτά τα έγγραφα, τα τελικά έγγραφα. Και το e-pitting έρχεται σε ένα περαιτέρω, μάλλον πιο ε, ύστερο στάδιο, έτσι ώστε να επικυρωθεί το έγγραφο κάθε φορά όταν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του. Θέλει κανείς άλλος? Ναι, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ πολύ για την ε, πρωτοβουλία. Εμείς ε, έχουμε στην Αυστρία κάνει ό,τι μπορούσαμε μέχρι τώρα για να μειώσουμε την σπατάλη χαρτιού. Εδώ βλέπω ότι έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε, επί παραδείγματι, για τις καρτέλες με τα ονόματα. Γιατί και αυτό σπατάλει χαρτιού ένα. Εν πάση θέλω να ρωτήσω το εξή. Βλέπω ότι δεν ε, έχω πρόσβαση ακόμα στην ε, βάση που έχω εγώ στον υπολογιστή μου από το iPad. Πώς μπορώ να το κάνω αυτό, γιατί δεν μπορώ να τα αξιοποιήσω. Είναι καλό να έχω τη δυνατότητα να βλέπω οποιαδήποτε έγγραφα. Απάντηση. Ναι, η εφαρμογή ίδια είναι προσβάσιμη, αν σας κατάλαβα καλά. Είναι ήδη προσβάσιμη η εφαρμογή. Οποιαδήποτε στιγμή, μέσα στη συνεδρίαση, πριν τη συνεδρίαση. Και ελπίζω να σας απάντησα. Μάρτιν. Δηλαδή εδώ μπορώ να έχω πρόσβαση. Πώς θα μπω στο σύστημα χωρίς να βρίσκομαι στον κύριο υπολογιστή. Μικρό Το μικρόφωνο σας παρακαλώ να κλείσετε. Ναι, θα χρειαστεί όμως να έχετε ένα ε, μηχάνημα, έτσι, ένα τάμπλετ ή ένα smartphone, ένα ευφυές τηλέφωνο. Η εφαρμογή μας ε, εξυπηρετεί οποιοδήποτε μηχάνημα και χρειάζεται να έχετε στα χέρια σαν ένα μηχάνημα, Αλλιώ δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση. It works, Όχι, εγώ νομίζω ότι δουλεύει. Παρακαλώ εσείς. Δεν ξέρω αν καταλάβατε ή όχι, πάντως το πρώτο τμήμα της ερώτησης του συναδέλφου δεν απαντήσατε. Ίσως είναι πρόβλημα συνεννόησης. Γιατί πρέπει να χαλάμε χαρτί κάθε φορά να έχουμε ας πούμε το χάρτη κάθε φορά των, ε, ε δογιο, των ε, ε, κάθε φορά να έχουμε χάρτη, να έχουμε boarding pass, κάρτες επιβίβασης, να τα δίνουμε και να τα ξαναδίνουμε. Ε, μπορούμε να κάνουμε ηλεκτρονικά την, ε, την δήλωση του ταξιδιού. Ε, το βράδυ ένα μικρό κοριτσάκι μου είπε θα μας σκοτώσετε, θα μας σκοτώσετε εσείς γιατί χωρίς δέντρα δεν θα έχουμε πια οξυγόνο εάν ε, συνεχίσουμε να καταναλώνουμε χαρτί με αυτούς τους ρυθμούς. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε ηλεκτρονικά τις δηλώσεις ταξιδίου μας. Yeah, sorry for that. Um, we are speaking here for, for a kind... Κοιτάξτε, μιλούμε εδώ για ένα κομμάτι της δουλειάς Καταλαβαίνω ότι πρέπει να καταβάλουμε και άλλες προσπάθειες για τα όσα έχουν να κάνουν με το χαρτί, αλλά εδώ μιλούμε για το μεγαλύτερο κομμάτι της κατανάλωσης του εγγράφου. Έχουμε εκτυπώσει 30 εκατομμύρια σελίδες πέρσι, για παράδειγμα. Είναι τεράστιο το νούμερο και προσπαθούμε να το μειώσουμε. Ορισμένες επιτροπές έχουν, λειτουργούν τελείως ηλεκτρονικά πλέον και δεν έχουν καθόλου εκτύπωση επί χάρτου. Είναι μια γενική πρωτοβουλία αυτή. Ένα μικρό βήμα κάνουμε, αν θέλετε, τώρα. Ένα πρώτο βήμα και Προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε όσο δυνατόν λιγότερα εκτυπωμένα ε, χαρτιά. Καταλαβαίνω απολύτως την ε, ανησυχία σας. Ε, Άλλη μια, στα γρήγορα. Υπόθηκε λοιπόν και θα ήθελα να μας εξηγήσετε λίγο περισσότερο το πώς μπορεί αυτή η εφαρμογή, αυτή είναι η ερώτηση νωρίτερα, πώς μπορεί αυτή η εφαρμογή να συνδέεται στον κύριο υπολογιστή που έχω στο γραφείο μου. Υπάρχει κάποιος σύνδεσμος, υπάρχει μια ποιοτική διαφορά ανάμεσα στο εάν θα χρησιμοποιήσω το ίντρανετ και έναν κοινό web browser, άλλες πληροφορίες θα λάβω. στο, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής. Τα βλέπω τα στοιχεία που μου λέτε, η μερίσια διάταξη, ε, φίλε, τα βλέπω. Υπάρχει κάποια διαφορά, λοιπόν. Και το πρόβλημα που έχω εγώ είναι ότι πολλές φορές ε, ψάχνοντας κάτι βρίσκω πολλές φορές το ίδιο πράγμα ότι δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των κατακόρυφων δομών του Κοινοβουλίου. Αυτό είναι το θέμα μας. Ναι, ευχαριστώ για την ερώτηση. Αυτό, αυτή η εφαρμογή, το e-meeting που βλέπετε, σας δείχνει τα ίδια έγγραφα, της ίδιας πληροφορίας με άλλο τρόπο. Εδώ επικεντρωνόμαστε μόνο στην πρακτική, στη συνεδρίαση. Έχουμε την ημερήσια διάταξη, τη σύνοδο, το, το όνομα της αίθουσας, όλα αυτά. Ένας διαφορετικό τρόπος να σας παρουσιάσει τα στοιχεία. Είναι αυτή η εφαρμογή. Ωστόσο, έχουμε υπόψη αυτή την εσωτερική εφαρμογή να την ενισχύσουμε με χαρακτηριστικά ειδικά της δουλειάς μας. Στην ιστοσελίδα της Επιτροπής σας θα δείτε μόνο δημόσια έγγραφα, προσβάσιμα στο κοινό. Εδώ μπορείτε να βρείτε και έγγραφα που είναι από συνεδριάσεις και ξενών των θυρών όπως των συντονιστών ή άλλες, εφόσον μπορέσουμε να συνδυάσουμε πάνω στοιχεία ασφάλειας επιπλέον. Προ το παρόν όμω είναι τα ίδια με αυτά που βλέπετε στην ιστοσελίδα. Ε, εμείς βεβαίως παρουσιάζοντας τους βουλευτές λαμβάνουμε και τι παρατηρήσει του και αυτέ είναι πολύ χρήσιμε, γι' αυτό σα παρακαλώ και εσάς. Ε, λοιπόν, άκουσα ένα σχόλιο από έναν βουλευτή που έλεγε Α, να ήμουν αφαιρεπίν σήμερα στην Επιτροπή των Μεταφορών και ταυτόχρονα υπήρχε μια άλλη επιτροπή στην οποία επίση είμαι μέλο και ήθελα να είμαι σε θέση να παρακολουθώ σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ημερήσια διάταξη της άλλης συνεδρίας, ώστε αν χρειαστεί να τρέξω να πάω στην άλλη συνεδρίαση. Άρα μπορούμε να έχουμε έναν κούρσορα εγκαταστημένο, ώστε να παρακολουθούμε παράλληλα κάποια άλλη επιτροπή. Mm. Μια ιδέα. Άλλος βουλευτής μας ρωτούσε αν μπορεί κατά τη διάρκεια της ε, συνεδρίασης να επικοινωνεί με instant messaging, ε, γιατί χρησιμοποιεί μόνο το SMS του τηλεφώνου αυτή τη στιγμή, με τον βοηθό, την βοηθό στο γραφείο για να ζητήσει κάτι που χρειάζεται κάτι τέτοιο, ένα instant messaging μπορεί να είναι μια λύση. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο, ευχαριστούμε για τι πληροφορίε σα και για τι απαντήσει που δώσατε. Πάμε στο επόμενο θέμα τη ημερήσια διάταξη, κατάσταση σε σχέση με του τριμερεί διαλόγου, καταρχά ε, σιδηροδρομικά, στατιστικές σιδηροδρομικές ιστορικών υδάτων και κλεισμένων των θυρών, ούτε Συμβούλιο, ούτε Επιτροπή θα είναι παρόντες, ούτε έτεροι Και γι' αυτό σας παρακαλώ να αποχωρήσουν όσοι δεν έχουν συνεργασία. Da kommt nicht, ne?